Herr Präsident! Bitte nehmen Sie. Ich erkläre die am 3. April unterbrochene Sitzung. Κυρίσω την επανάληψη της Συνόδου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που είχε διακοπεί στις 3 Απριλίου. Κυρίες και κύριοι, νομίζω ότι όλοι είμαστε ιδιαίτερα ανήσυχοι. Είμαστε ιδιαίτερα ανήσυχοι εξαιτία των εξελίξεων που προχωρούν όλο πιο γρήγορα και είναι και όλο πιο δύσκολε στην Ουκρανία. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πάντως στην μεγάλη του πλειοψηφία επιμένει για την εδαφική ακεραιότητα και την κυριαρχία στην Ουκρανία. Σε πολλά ψηφίσματά μας έχουμε ήδη πει ποια είναι η άποψή μας. Εξάλλου θα το συζητήσουμε και αυτή τη βδομάδα.